Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αρχίζουν οι ψηφοφορίες. Θα ψηφίσουμε πρώτα, με βάση την απλουστευμένη διαδικασία, την έκθεση του κυρίου Μαστάλκα με θέμα της συγχωνεύσης των ανωνύμων εταιριών. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Se cierra Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η έκθεση. Δεύτερο θέμα, σύσταση Αλμπερτίνη. Πρωτόκολλο Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιορδανία. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Έκθεση Κοχ. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών. Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, ζήτησε το λόγο ο εισηγητής ο κύριος Κοχ. Σας ακούμε κύριε Κοχ. Αγαπητοί συνάδελφοι, με την έγκριση της εκθεσισμού συνδεχόμετα και μία συμφωνία δεχόμεθα την προσαρμογή 47 συμφωνιών ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ε, τις, ε, τις χώρες της Αφρικανικής Ένωσης. Βεβαίως αυτό θα οδηγήσει στο να μην υπάρχουν διακρίσεις και γραφειοτικές διαδικασίες και παρακαλώ που να συμφωνήσετε σε αυτή τη συμφωνία με τη Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. Σε δεύτερη ανάγνωση εξετάζουμε τη θέση του Συμβουλίου για τους εναρμονισμένους όρους εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Η συγγήτρια είναι η κυρία Στήλερ και ψηφίζουμε πρώτα το πρώτο σύνολο τροπολογιών, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εγκρίνεται η θέση του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από το Κοινοβούλιο. Ψηφίζουμε τώρα την έκθεση Στρίφλερ για την Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη περί ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν έχουν κατατεθεί τροπολογίες, αλλά έχουμε πολλές ψηφοφορίες κατά τμήματα ή ξεχωριστές. Ψηφίσουμε πρώτα σε δύο τμήματα την παράγραφο 5. Πρώτο τμήμα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφο 9. Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Σε Τέλος. Εγκρίνεται η Παράγραφο 9. Παράγραφος 13. Σε δύο τμήματα. Και τα δύο θα τα ψηφίσουμε ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία, ονομαστική κλίση για το πρώτο τμήμα. Τέλος. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα της, της παραγράφου 13. Παράγραφος 31. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Παράγραφος 32. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται και αυτή. Παράγραφος 33. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 35. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. Παράγραφος 39. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη σε. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα της αιτιολογικής σκέψης σε γάμο. Σε θύαρα, Τέλος. Δεύτερο τμήμα, το δεύτερο τμήμα της αιτιολογικής σκέψης σε εγκρίνεται με μία ψηφοδιαφορά, διαφορά οριακά. Τρίτο τμήμα τώρα της αιτιολογικής σκέψης σε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος και πάλι για το τρίτο τμήμα της αιτιολογικής σκέψης C. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Το τρίτο τμήμα εγκρίθηκε με 10 ψήφους διαφορά αυτή τη φορά. Αιτιολογική σκέψη G. Δύο τμήματα. Ποιο είναι υπέρ του πρώτου τμήματο. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε τώρα το σύνολο της πρόταση. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Παίρναμε τώρα στην έκθεση Σαρμπού για τη Γεωργία ως στρατηγικό τομέα στο πλαίσιο της επιστημιστικής ασφάλειας. Δεν έχουν υποβληθεί τροπολογίες, αλλά και πάλι θα ψηφίσουμε ξεχωριστά ορισμένες παραγράφους. Αρχής γενομένης από τις παραγράφο 8, που θα την ψηφίσουμε σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση για το πρώτο τμήμα της παραγράφου 9. Πολύ ωραία. Ας το ελέγξουμε. Πρώτο τμήμα τη παραγράφου 9. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος. Εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. 300 ψήφους. Και. Δεύτερο τμήμα τώρα της 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 14. Σε τρία τμήματα, ονομαστικές ψηφοφορίες και τις τρεις φορές. Για το πρώτο τμήμα έρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα με σαφή διαφορά. Δεύτερο τμήμα, Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Τρίτο τμήμα τώρα, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Το τρίτο τμήμα απορρίπτεται. Παράγραφος 24 σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 27 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Vamos a eh, se, cierra la votación. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα της 27 και τώρα τρίτο τμήμα της ε, παραγράφου 27. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 29, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 30, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 31, ποιος είναι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 36, σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σε δύο τμήματα, 45, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για το πρώτο τμήμα της παραγράφου 45 Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα της 45. Σε Τέλος. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Τροπολο... Ε, παράγραφος 50 σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Παράγραφος 51 σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη π. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την αιτιολογική σκέψη π. Τέλος ψηφοφορίας. Η αιτιολογική σκέψη π Απορρίπτεται η σοπαλία. Όχι, δι, διορθώνει ο πρόεδρο. Εγκρίνεται η αιτιολογική σκέψη π. Vamos Έχετε το λόγο, κύριε Νέα, Κύριε Πρόεδρε, έχουμε πρόβλημα εδώ. Και τα δύο μηχανήματά μας δεν λειτουργήσαν. Bueno, pues le enviamos un técnico. Bueno, Ωραία, θα σας στείλουμε τεχνικό. Sobre la votación del Στην αιτιολογική σκέψη, πει λατινικό, έχουμε ισοψηφία. Αν ήταν τροπολογία, που να τροποποιεί το κείμενο δηλαδή, η τροπολογία θα το. Τι συμβαίνει τώρα. Επειδή δεν πρόκειται για τροπολογία, αλλά για αιτιολογική σκέψη του κειμένου, στην περίπτωση αυτή, με ενημερώνουν οι υπηρεσίες και τις πιστεύω ότι στην περίπτωση αυτή η ισοψηφία ισοδυναμεί με έγκριση του κειμένου. Οπότε η αιτιολογική σκέψη πει λατινικό εγκρίνεται. Και θα ψηφίσουμε το σύνολο της πρότασης. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ και ακολουθούν επεξηγήσεις ψήφου. Πού Good. Empezamos por el informe de la señora Stiller. Αρχίζουμε από τη λέξη κυρία Στάιλερ.